θα μπορέσει να ισχύσει και να κοιτάξουμε να μεταρρυθμίσουμε αυτή τη διαδικασία της απαλλαγής. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, πρωτού προχωρήσουμε στην, στον κατάλογο των ομιλητών θα ήθελα ε, εδώ να κάνω ορισμένες διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 ε, ε, του εσωτερικού κανονισμού για ορισμένες προθεσμίες. Υπάρχουν τέσσερις διορθώσεις τις οποίες πρέπει να διαβάσω. Ευχαριστώ και πρόκειται καταρχήν για τις αρμόδιες επιτροπές διότι οι ε, ε, επιτροπές έχουν δώσει διορθώσεις στο Προεδρείο καταρχήν για την έκθεση η οποία εξετάστηκε στις 24 Νοεμβρίου του 2010 για τον περιορισμό χρήσεως επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρονικά όργανα Δεύτερον, σχετικά με την έκθεση που αποφασίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου σχετικά με την οδηγία για την αλλαγή της οδηγίας 2001-300 ε, ε, για τα φάρμακα ε, και για παραποιήσεις που γίνονται στην αλυσίδα της διαθέσης στο Τρίτον, για μία έκθεση ε, σχετικά με μία απόφαση του Συμβουλίου ε, ε, στην ε, τροποποίηση μίας οδηγίας για τα δικαιώματα του τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα και τρίτον εις την αλλαγή της οδηγίας για τους διαχειριστές των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων και της της ε, ε, αρμοδίας αποφάσεως και των κανονισμών που άπτονται του θέματος αυτού. Σύμφωνα με ε, τον εσωτερικό κανονισμό θεωρούνται ότι οι διορθώσεις αυτές θα ισχύσουν εφόσον ε, εντός 48 ωρών δεν έχει ζητηθεί από τουλάχιστον 40 ε, βουλευτές να υπάρξει νέα ψηφοφορία επί το θέματος. Και τώρα προχωράμε στον κατάλογο των ομιλητών και δίνω το λόγο